Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Χαιρετίζω την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιεν, καθώς επίσης και την Υπουργό εκπρόσωπο της Προεδρίας ε, του Συμβουλίου. Η μερίσια διάταξη προβλέπει ω πρώτο θέμα τι δηλώσει του Συμβουλίου και τη Επιτροπή σχετικά με την προτινόμενη εντολή για διαπραγματεύσει σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με τον Ηνωμένο Βασίλειο τη Μεγάλης Βρετανία και τη Βόρειας Ιρλανδίας. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω ε, εξ ονόματο Συμβουλίου στην Υπουργό Μπέρνετ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης και την αποχώρηση λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάνε νέες διαπραγματεύσεις. Προκειμένου αυτές να λάβουν χώρα θα πρέπει να υπάρχει μια εντολή προς τον διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει σωστή βάση για την εντολή αυτή. Ω προ αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να σε εκθέσω κάποιε βασικέ σκέψει όσον αφορά την προετοιμασία αυτή τη εντολή για διαπραγματεύσει. Καταρχά, όσον αφορά την περιεκτική αυτή εντολή που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πεδίο εφαρμογή διαπραγματεύσεων αυτών ιδιαίτερα ευρύ. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθυστερήσουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων αυτών. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να ξεκινήσει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει και να εγκριθεί η προτινόμενη εντολή για διαπραγματεύσει, και αυτό προβλέπεται να γίνει στι 25 Φεβρουαρίου στι σχετικέ συνεδρίε του Συμβουλίου. Και αυτό ουσιαστικά σχετίζεται και με την απόφαση του Μπόρι Τζόνσον να μην επεκταθεί πέρα από την 31η Δεκεμβρίου η μεταβατική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πολλέ διαπραγματεύσει να κινηθούν παράλληλα. Αυτή η εντολή λοιπόν, μιλάμε για εντολή για διαπραγματεύσει και όχι για τελική έκβαση διαπραγματεύσεων. Και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να γνωρίσουμε ακριβώ πού θα καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε, ποιε ήταν τελικέ προσφορέ, ποιε θα πρέπει να είναι οι παραχωρήσει οι οποίε θα πρέπει να λάβουν χώρα θα πρέπει να έχουμε επίση την απαραίτητη ευελιξία. Επίση, και εδώ πέρα αναφέρομαι και στο ζήτημα τη ενότητα, καθώ επίση και του περιορισμένου χρόνου, μια πολύ περιοριστική εντολή για διαπραγματεύσει θα πετούσε περισσότερο χρόνο προκειμένου να καταφέρουμε να γεφυρώσουμε αποκλήσει και να προωθήσουμε συγκεκριμένε προτεραιότητε. Ανταυτού, θα πρέπει να προωθήσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχουμε μια έκβαση η οποία είναι ανισότιμη και συμφέρουσα για όλα τα κράτη-μέλη και του πολίτε του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να δούμε ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του πρόθεση της κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει την ελεύθερη κυκλοφορία και αυτό προφανώς θα στραφεί κατά των δικαιωμάτων κινητικότητα και κυκλοφορίας των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό επίση να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και εν γέννη στο εμπόριο. Επί τη ουσία, όσον αφορά την προτινόμενη αυτή εντολή για διαπραγματεύσει και του διάφορου τομεί που θα πρέπει προφανώ να καλύψουμε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, μάλλον συμφωνούμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, όπω φαίνεται και από το σχέδιο ψηφίσματό σα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ένα καλό επίπεδο φιλοδοξία σε σχέση με τη σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλε χώρε. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε στον Μένο Βασίλειο τα ίδια ωφέλη που θα είχε όπω όταν ήταν κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τι κόκκινε γραμμέ που έχει θέσει βέβαια. Α δούμε κάποια οριζόντια ζητήματα τη εταιρική σχέση, τη διακυβέρνηση, καθώ επίση και του ισότιμου επίπεδου ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να προσφέρουμε μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ελεύθερη πρόσβαση στο εμπόριο, αλλά αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να στραφεί κατά τη ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ή των ε, κανόνων κρατικών ε, ενισχύσεων. Και βέβαια στην εταιρική αυτή σχέση θα πρέπει να έχουμε πολλέ διατάξει όσον αφορά το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού βασιζόμενοι σε πολύ ψηλά πρότυπα. Και βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λαμβάνοντα υπόψη την πρόθεση του Βασιλείου να αποκλίνει και να από την, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια αυτό σχετίζεται και με το ζήτημα της αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών, καθώς επίσης και με το ζήτημα των αποζημιώσεων και της επιβολής των νομοθεσιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ισότιμους κανονισμούς, οι οποίοι να μπορούν όμως να εφαρμόζονται. Πρώτα ολοκληρώσω δύο σημαντικέ παρατηρήσει. Πρώτον, μολονότι όλοι γνωρίζουμε ότι η γραμμή τη Βρετανική κυβέρνηση είναι να θέσει ένα τέλο στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, η μελλοντική σχέση την οποία θα πραγματευτούμε θα πρέπει να είναι αρκετά φιλόδοξη όσον αφορά το ζήτημα της κινητικότητας. Δεύτερον, και αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη παρατήρηση που έκανα, οι διαπραγματεύσεις αυτές θα απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης για μία ακόμη φορά λοιπόν θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια όλων των μελλοντικών διαπραγματεύσεων θα έχουμε όλοι ένα κοινό συμφέρον να έχουμε μια καλή συνεργασία με τον Ηνωμένο Βασίλειο καθ' όλη αυτή τη διάρκεια της περίοδου αποχώρησης. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Τώρα το λόγο έχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Φόντερ Λάιεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες αποχαιρετήσαμε τους Βρετανούς συναδέλφους ε, τραγουδώντας τον αποχαιρετιστήριο αυτό ύμνο. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή, πολύ δυνατή στιγμή εδώ στο Κοινοβούλιο και μια στιγμή που γιορτάσαμε τις παλιές καλές στιγμές. Και ήταν πάρα πολύ ευγενική αυτή η χειρονομία. Ε, έκτοτε θέτουμε τα θεμέλια ε, για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές με την υψηλότερη δυνατή φιλοδοξία. Γιατί δεν θα πρέπει να συμβιβαστούμε με λιγότερα, ούτε οι Βρετανοί ούτε εμεί. Ο, ο Πρωθυπουργό Τζόνσον είχε πει στο Greenwich πρόσφατα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και παραθέτω θα είναι ε, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής ελευθέρου εμπορίου. Τέλος της παράθεσης. Ειλικρινά, αυτό είναι μουσική στα αυτιά μας. Γιατί τη στιγμή όπου το σύστημα εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες ε, δοκιμάζεται, χρειαζόμαστε εταίρους έτσι ώστε το σύστημα να γίνει και πιο δίκαιο και πιο ισχυρό. Μα γι' αυτό έχουν αγωνιστεί οι Ευρωπαίοι όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύστημα εμπορίου που να είναι από τη μια ανοιχτό, αλλά από την άλλη και δίκαιο. Γιατί? Τι κάνουν οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου? Θα πρέπει να αντικαθιστούν την ανασφάλεια από ένα σύστημα κανόνων αξιόπιστων. Νέες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα ε, είναι το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο υπέρ των ανθρώπων. Αυτή είναι η λογική πίσω από τις δικές μας ε, ε, σχέσεις και συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, ας πούμε, με την Ιαπωνία ή τον Καναδά. Δεν αυξάνουν μόνο τις συναλλαγές μας σε εμπορεύματα, υπηρεσίες, ανθρώπους και ιδέες που το κάνουν και αυτό, αλλά ανεβάζουν τα πρότυπα ε, και για τα εργασιακά ζητήματα, τις συνθήκες εργασίας και τα περιβαλλοντικά. Και αυτό ζητούμε και από τους Ιάπωνες ή τους Καναδούς φίλους μας. Και χαίρονται που συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας έτσι ώστε να φέρουμε περισσότερη δικαιοσύνη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Χαίρονται που μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εκείνοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ειλικρινά στο σημερινό κόσμο μετράει το μέγεθος. Και εμείς έχουμε μια ενιαία αγορά 440 εκατομμυρίων πολιτών. Αυτό που μόλις σας περιέγραψα είναι η δική μας φιλοδοξία για τις συμφωνίες ελευθερου με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή τη στιγμή συμφωνήσουμε για την πολιτική δήλωση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε στόχο για μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις για τις συναλλαγές σε όλα τα αγαθά. Κάτι που ουδέποτε στο παρελθόν δεν είχαμε προσφέρει σε κανέναν. Ένα νέο μοντέλο εμπορίου μοναδική φιλοδοξία για πρόσβαση στην ελεύθερη εσωτερική αγορά, αλλά φυσικά αυτό σημαίνει και αμοιβαιότητα με εγγύσει για δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό, για την προστασία των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και καταναλωτικών προτύπων. Αυτό είναι ε, ίση κανόνε παιχνιδιού. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε όλα τα διαφορετικά μοντέλα συμφωνίας εμπορίου. Όμως, οτιδήποτε και αν επιλέξει κανείς, Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ένα κοινό. Δεν συνοδεύονται απλώς από δικαιώματα αλλά και από υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές. Παράδειγμα, ας δανειστούμε το μοντέλο του Καναδά στο οποίο είχε αναφερθεί και ο Πρωθυπουργό Τζόνσον. Βεβαίω, η συμφωνία μα με τον Καναδά καταργεί του δασμού σε πάρα πολλά προϊόντα, αλλά όχι σε όλα. Και φυσικά η συμφωνία μας με τον Καναδά καταργεί τις περισσότερες ποσοστώσεις, αλλά σίγουρα όχι όλες. Ας πούμε για το γλυκό αραβόσιτο και ε, το βόλιο κρέας. Φυσικά έχουμε ακόμα τις δικές μας ε, αρχές και προδιαγραφές και πρότυπα που πρέπει να γίνονται σεβαστά. Και ειλικρινά ξεπλάγει λίγο όταν άκουσα τον Πρωθυπουργό του Ρωμανού Βασιλείου να ομιλεί για το αυστραλιανό μοντέλο. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι η Αυστραλία είναι ισχυρό εταίρο και στη δική μας κατεύθυνση. Αλλά εμεί δεν έχουμε εμπορική συμφωνία με την Αυστραλία. Ε, έχουμε εμπόριο βάσει των κανόνων του ΠΟΕ. Και αν αυτή είναι η επιλογή των Βρετανών, πολύ ωραία και δεν το αμφισβητούμε. Αλλά Τώρα ε, συζητούμε με τους ε, Αυστραλούς για μια νέα συμφωνία. Φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συμβιβαστεί με λιγότερα, αλλά ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτή η φιλοδοξία μας. Και στο Greenwich η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι μια καλή ενθαρρυντική αφετηρία. Θύμισε όλα τα επιτεύγματα του Ηνωμένου Βασιλείου στην κοινωνική προστασία, στην κλιματική δράση, στους αγώνες ανταγωνισμού και το συγχαίρω του Ηνωμένου για όλα αυτά. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να ε, ρίξουμε την κοινωνική προστασία, να είμαστε χλιαροί ε, στην κλιματική δράση. Δεν είναι η ώρα να μειώσουμε ε, τους κανόνες ανταγωνισμού. Έχω ένιωσα φιλοδοξία στην ομιλία του Μπόρις Τζόνσον για τον κατώτατο μισθό, για πληρωμένη γονική άδεια. Άκουσα και φιλοδοξία για να μειωθούν οι εκπομπές διοξοδίου του άνθρακα φιλοδοξία για ανταγωνισμό των επιχειρήσεών μας σε πλήρη δικαιοσύνη. Και εμεί το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, α το συμφωνήσουμε επίσημα ότι είναι αυτή η στόχη μα και μπορεί να απογειωθεί ο δυναμικό ανταγωνισμό προ όφελο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου. Λέγω λοιπόν στου Βρετανού φίλου μα, είναι προ το κοινό μα συμφέρον και κυρίω αυτό θα συνάδει με τις αξίες που μοιραζόμαστε, τις αξίες του ανοιχτού πνεύματος της δικαιοσύνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του ελεύθερου επιχειρήν και αυτά. Δεν είναι μόνο αξίες του παλιού καλού καιρού. Είναι αϊθαλείς αξίες αυτές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ενημερώνω ότι η Task Force είναι έτοιμη να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Πανέτοιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστούμε Πρόεδρε. Ας ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, ξεκινώντας από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο κύριος Μακάλιστερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Μινουτι. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι, το ψήφισμα για την εντολή διαπραγμάτευση που συζητούμε σήμερα το πρωί είναι το πρώτο, η πρώτη απόδειξη ε, του έργου που έχει κάνει αυτή η νέα ομάδα συντονισμού για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω ως πρόεδρος να ευχαριστήσω όλα τα μέλη αυτής της ομάδας, τι πολιτικές ομάδες για τις συνεισφορέ τους σε μια πάρα, πάρα πολύ μικρή χρονική περίοδο που μεσολάβησε. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι καλό, έχουμε ένα ισορροπημένο ψήφισμα Μόλις 9 μέρες αφού ο Μισελ Μπαρνιέ παρουσίασε το σχέδιο εντολής διαπραγμάτευσης της ε, Κομισιόν. Επικεντρωνόμαστε στο περιεχόμενο και στην αρχιτεκτονική των μελλοντικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να αναδείξω τρεις βασικές αρχές που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές. Πρώτον, η ακαιρεότητα και η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Τελωνιακή Ένωση και οι τέσσερι ελευθερίες πρέπει να διατηρηθούν. Δεύτερον, μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα και ωφέλη όπως αυτά που έχει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, η ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε έναν αγώνα προς τα κάτω. Όπως ε, ε, είπε και η κυρία Φόντερ Λάιεν, μαζί με τους Βρετανούς φίλους μας πρέπει να στοχεύσουμε σε μια εταιρική σχέση η οποία θα υπερβαίνει το εμπόριο και που δεν θα είναι προ, ε, από άποψη εύρους. Αλληλεία, προστασία προσωπικών δεδομένων, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ασφάλεια. Θέλουμε να σχεδιάσουμε μια νέα εταιρική σχέση χωρίς δασμούς, χωρίς ποσοστώσεις και χωρίς dumping. Όμως, μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ε, αποτελέσει ένα ε, ε, ε, ένα ε, μπούσουλα για εμπόριο χωρίς καθόλου τριβές. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών και το πρωτόκολλο του, που έχει υπογραφεί για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ε, ήδη στην πρώτη συνάντηση της ομάδας συντονισμού ο Μισελ Μπανιέ μας ε, ε, εγγυήθηκε ότι θα ενημερώνεται διαρκώς το Κοινοβούλιο για όλα τα βήματα και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται. Κυρία Γκαρσία Πέρετς, τώρα έχει το λόγο ξενόματος των σοσιαλιστών. Τρεις ή λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματο της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα την ομάδα του κυρίου Μπαρνιέ για τις προσπάθειές σας για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών έτσι ώστε να διαπραγματευτούμε το πλαίσιο των μελλοντικών μας σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτό που πρόκειται να εγκρίνουμε, στέλνουμε ένα στεναρό μήνυμα. Η φιλοδοξία για τις μελλοντικέ σχέσει θα εξαρτηθεί από τη βούληση της κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ευθυγραμμιστεί στα κοινωνικά, εργασιακά, φορολογικά και περιβαλλοντικά πρότυπα την 1η Φεβρουαρίου και τυπικά το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε τρίτη χώρα και έχασε όλα τα πολιτικά του δικαιώματα. Σε όλα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα όμως μέχρι να τελειώσει η μεταβατική περίοδος. να αλλαξει τιποτα ομω μεχρι να τελειωσει η μεταβατικη περιοδος εχουμε 11 μήνε για να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία περίπλοκη που θα καθορίζει τι μελλοντικέ μα σχέσει. Εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, δεν θα υπάρχουν πλέον εκτίματα τύπου κράτους μέλους. Εμείς θέλουμε να υπάρχει συνολική συμφωνία. Αλλά όσο περισσότερα εμπόδια ορθώνει το Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνησή του, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ε, καταλήξουμε σε φιλόδοξη συμφωνία. Από την άλλη, αν έχει την πρόθεση να παραμείνει θεμητός ανταγωνιστής και έντιμος, εμείς θα τους προσφέρουμε μια συμφωνία που θα εγγυάται την ευημερία εκατέρωθεν της μάνχης. Και για να γίνει αυτό ναι στην κατάργηση δασμών, ναι στις ποσοστώσεις για όλα τα αγαθά που ε, μπαίνουν στην εσωτερική αγορά αλλά και για τις υπηρεσίες. Αν θέλουμε να είναι όμως πραγματικά τα ωφέλη, χρειαζόμαστε μια ε, ε, εταιρική σχέση στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια και άμυνα, στην παγκόσμια τάξη, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στην αλία και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Όμως δεν θα πρέπει να γίνει ε, με οποιοδήποτε τίμημα αυτό. Θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να εγγυηθεί θεμητό ανταγωνισμό. Να ε, υπάρχει εγγυημένη πρόσβαση του αλευτικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατά της και επίσης να τηρεί και να εφαρμόζει τις αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και επίσης να σεβαστεί τα όσα ισχύουν για το Γιβραλτάρ όπως ε, κυρώθηκε στις κατευθυντήριες γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ε, επιτυχία μας θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε αυτό που μέχρι τώρα ήταν το καλύτερο όπλο μας, την ενότητα. Μοναδικό συνομιλητή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την τελική συνένεση έχει λόγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο έτσι θα μπορέσει μέχρι, τη μέχρι τώρα ενότητα να τη διατηρήσει. Έχουμε καταφέρει ε, την ακαιρεότητα των τεσσάρων ελευθεριών τη Τελωνιακή Ένωση ε, και την ελεύθερη κυκλοφορία φυσικά των πολιτών. Α μην ξεχνάμε ότι ε, βασιζόμαστε σε μία δέσμευση με συγκεκριμένε αξίε που είναι ακριβώ αντίθετε από εκείνε που ακούμε από κάποιου Βρετανού ηγέτε που εμφορούνται ε, από εθνικισμό και ε, μία λανθασμένη ιδέα ανωτερότητας. Έχουμε την ευθύνη τώρα να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που μας επέτρεψαν το ευρωπαϊκό μας εγχείρημα να προχωρήσει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος τώρα της ομάδας Renew Europe, η κυρία Λουαζό έχει το λόγο για δυόμιση λεπτά το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένοι ενδεχομένω να βλέπουν εδώ πέρα μια αντίφαση που θα έκανε τι διαπραγματεύσει μεταξύ ημών ακόμα πιο δύσκολε. Εγώ νομίζω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί εμεί ουσιαστικά σεβόμαστε την επιλογή των Βρετανών πολιτών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά από την ενιαία αγορά και την Τελωνιακή Ένωση. Πρόκειται για μια ριζοσπαστική επιλογή την οποία εμεί σεβόμαστε. Προφανώ υπάρχουν συνέπειε τι οποίε δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και θα διαμορφώσουμε σε σαφώ τη μελλοντική μα σχέση. Βέβαια, χρειαζόμαστε μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση και για την, το ίδιο Βασίλειο. Είμαστε άμεσοι γείτονε και είμαστε ο βασικό εταίρο του Λονδίνου όσον αφορά τι εμπορικέ αλλά και τι ανθρώπινε σχέσει. Ε, έχουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία πραγματικά θα πρέπει να σεβαστούμε. Και βέβαια έχουμε μια τεράστια πρόκληση την οποία από κοινού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική αλλαγή, τρομοκρατία, επιθέσει ε, στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι απλώνονται και δεν γνωρίζουν σύνορα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πολεμήσουμε τα φαινόμενα αυτά με νέα μέσα από κοινού, και διαφορετικά θα χάσουμε και οι δύο, και οι δύο πλευρέ. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βιώσιμη, ισχυρή εταιρική σχέση με το Μέντο Βασίλειο και είμαστε παράλληλα πεπισμένοι ότι ε, το Brexit σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο τη μεταξύ μόνη σχέση. Έχουμε υψηλά πρότυπα για να προστατεύσουμε του καταναλωτέ, για να προστατεύουμε του εργαζόμενου, για να προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών μα. Και προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύουμε τελικά ακόμα και τον ίδιο τον πλανήτη μα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε υποχωρήσει και εκχωρήσει τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε μάχη και θα συνεχίσουμε για τα ζητήματα αυτά να δίνουμε μάχη. Η προτινόμενη το λέγεται πραγματεύσιμο το Βασίλειο καταδεικνύει ακριβώς ε, την δυναμική αυτή σχέση την οποία θέλουμε να έχουμε με τη χώρα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να καλύψουμε στο πεδίο εφαρμογή πολλού διαφορετικού τομεί. Ζητάμε λοιπόν και από το Μένο Βασίλειο να καταφέρει πραγματικά να αποκριθεί στι ε, υποχρεώσει που του ζητάμε, όπω γίνεται ακριβώ και με άλλε χώρε με τι οποίε συνεργαζόμαστε γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη, είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε εμά, πολύ πιο δεσμευμένη, ε, συνδεδεμένη μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό το Brexit να μην χωρίσει και δεν μπορεί να χωρίσει τον κοινό πολιτισμό που έχουμε, καθώς επίσης και την ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή οικοδόμηση, την οποία διαμορφώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Εξ ονόματος των, ε, της ομάδας ID, ο κύριος Κόφοντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Οι Βρετανοί είναι και θα παραμείνουν στενοί φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι. Εγώ θέλω μια συμφωνία με τους Βρετανούς η οποία θα σέβεται και θα ανταποκρίνεται στις ε, απαιτήσεις των Βρετανών ώστε να ε, αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποιος μπορεί να μπαίνει για παράδειγμα στη χώρα τους αλλά ε, και όσον αφορά τις υπηρεσίες. Θέλουμε όμως μια στενή συνεργασία με τους Βρετανούς στο εμπόριο. Είναι σημαντικό για τη χώρα μου, τη Δανία, να συνεχίσουμε να έχουμε δυνατότητα να έχουμε μια πολύ στενή εταιρική σχέση εμπορική με την Βρετανία. Η Δανία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς γιατί θέλαμε εμπορικές σχέσεις με την Βρετανία. Όταν ε, οι Βρετανοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν, είπαν ότι δεν εγκαταλείπουμε τον κόσμο ή την Ευρώπη, απλώ το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και αυτό είναι ένα στόχο θε, Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους Βρετανού, όπου το Brexit θα αποτελέσει μια αφορμή για να έχουμε μια συνεχιζόμενη στενή σχέση με του ε, Βρετανού, η οποία θα εξυπηρετεί τι κοινέ μα αξίε μια συνεργασία στη βάση της κοινή λογικής για το κοινό μας συμφέρον και όχι ε, και σε αντίθεση μάλλον με, τον, με την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που πολλές φορές υποστηρίζεται πολλές φορές και σε αυτό το κοινοβούλιο. Πρόεδρος των Πρασίνων κύριο Λάμπερς, αγαπητοί συνάδελφοι πρώτον. Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται γεωγραφικά. Επομένω, θα πρέπει να έχουμε στενέ και φιλικέ σχέσει, όσο το δυνατόν πιο φιλικέ και πιο στενέ. Δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διέπεται από έναν εθνικισμό. Εμείς βρίσκουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο πάρα πολλούς ε, φίλους. Όσον αφορά τώρα την εμπορική πολιτική, φιλοδοξία Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου είναι αντιφατικέ, ανταγωνιστικέ. Θέλουν να έχουν πρόσβαση στη δική μας την αγορά, αλλά δεν θέλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένου ευρωπαϊκούς κανόνες και περιορισμούς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε δημιουργικοί στον τομέα αυτό, τον εμπορικό, και θα ήθελα εδώ να δώσω κάποιες εξηγήσει. Εν γέννη, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών χρησιμοποιούνται από τις κεφαλουικές αγορές πολλέ φορέ για να δημιουργήσουν ένα κατώτατο επίπεδο όσον αφορά τι εργασιακέ, φορολογικέ, περιβαλλοντικέ σχέσει και πρότυπα. Εμεί εδώ πέρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε συμφωνία Ελεύθερο συναλλαγών με τον Μανέο Βασίλειο για να κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Επί του παρόντο, η νομοθεσία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μανδέου Βασιλείου είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένε όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνισμού, αλλά όχι όλα τα ζητήματα. Όσον αφορά την προστασία τη προσωπική ζωή, όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα, το Ευρωπαϊκή... η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο φιλόδοξη Βασίλειο. Υπάρχουν όμω άλλοι τομεί όπου το νομόνιο Βασίλειο έχει πιο φιλόδοξα πρότυπα. Για παράδειγμα, στον περιβαλλοντικό τομέα ή στον τομέα τη τραπεζική ρύθμιση. Θα μπορούσαμε λοιπόν στη νέα αυτή συμφωνία να έχουμε ένα κανόνα σύμφωνα με τον οποίο οι δύο εταίροι θα έπρεπε να εφαρμόσουν τα πρότυπα τα πιο υψηλά από τις δύο πλευρές, τα πιο φιλόδοξα πιο φιλόδοξα είναι αυτά τα οποία προστατεύονται περισσότερο την υγεία, την ιδιωτική ζωή, τι εργασιακέ συνθήκε, τι αμοιβέ. Αυτά προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία αναβάθμιση των προτύπων αυτών μέσω τη συνεργασία αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση και του Μένου Βασιλείου. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, θα μου πείτε ποτέ στο παρελθόν. Μα ακριβώ αυτή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε και ουσιαστικά αυτό συνάδει και με τη συμφωνία αυτή την οποία θα ψηφίσουμε σε λίγο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Ο κύριος Σέπινγκ τώρα εξ ονόματος ομάδας ECR για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ο χρόνος ε, μας πιέζει για την ε, σύναψη συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με την ε, Βρετανία. Οι διαπραγματεύσει στην ουσία θα πρέπει να βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων. Υπάρχει και μια νοοτροπία όμως η οποία θα πρέπει να διέπει τι σχέσει μας και στι δύο πλευρές της μάχης. Κάθε γραφειοκρατία επιμένει στις δικές της, στους δικούς κανόνες αποδίδοντας ιερό χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη ε, οι αρχές που διέπουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωση πολύ συχνά προσωμιάζουν με εκείνες που ε, ε, διέπουν παλιότερα στο παρελθόν μάλλον την Κινέζικη Αυτοκρατορία. Η Βρετανία είναι διαφορετική. Ε, οι Βρετανοί πολλές φορές έχουν την αίσθηση ότι ακόμη θέλουν να είναι, ε, ότι είναι ακόμη αυτοκρατορία και δεν θέλουν ε, να τους επιβάλλονται κανόνες απ' έξω. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε ε, απογοητευμένοι. Έγινε το Brexit και πρέπει πρώτα στην πρώτη θέση να θέσουμε τους πολίτες μας. Τελείωσε αυτό. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε σε απτά αποτελέσματα και όχι σε αρνητικά συναισθήματα. Η τρέχουσα Βρετανική κυβέρνηση είναι η πιο σταθερή στην Δυτική Ευρώπη. Με μεγάλη μεγάλη πλειοψηφία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ποιο άλλο θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Όμω πρέπει να μην υπερεκτιμούμε του κανόνε που μπορεί να λειτουργήσαν για αιώνε, αλλά δεν λειτουργούν πλέον. Μόνο με, αυτή την, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Και αυτό το ψήφισμα είναι μια καλή αφετηρία για τι διαπραγματεύσει. Κύριε Μπαρνιέ, είστε εμπειρό διαπραγματεύτη. και ελπίζω ότι θα καταφέρετε να πείσετε τους Βρετανούς εταίρου μα που μα χωρίζουν μόλις 30 χιλιόμετρα αλλά τελικά και δύο κόσμοι. Ο πρόεδρος Σίντερβαν τώρα εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Συνοδική Αριστερά για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στι διαπραγματεύσει για τι μελλοντικέ σχέσει Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ένωση Περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι μόνο οι μελλοντικέ οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, πώς αυτές θα διαμορφωθούν, αλλά πολλά περισσότερα. Πρόκειται για το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε. Δεν είναι αυτό το τέλος του παιχνιδιού, ούτε οι ερχόμενοι 11 μήνες, αλλά μπορεί να είναι αποφασιστική για να αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα κρίνει επίσης και το κατά πόσο ε, είναι πιο ελκυστικό μοντέλο ανάπτυξης το να είσαι μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά λοιπόν δεν είναι η οικονομία αγαπητοί συνάδελφοι το καθοριστικό, αλλά οι πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ο λεγόμενος απλός κόσμος που αποφασίζει ποιο θα είναι το πιο ελκυστικό μοντέλο ανάπτυξη. Αυτό μας έχει διδάξει το Brexit. Η εντολή την οποία σήμερα συζητούμε θα πρέπει να σέβεται λοιπόν τα συμφέροντα του λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου και να τα φέρει στο κέντρο. Η ε, ομάδα μου καλωσορίζει ε, τις σαφεί δηλώσει για την προστασία από το φορολογικό ε, dumping, για τα κοινωνικά, για τα περιβαλλοντικά, για τα κατανοητικά. Κανένα δεν θέλει dumping και τελικά δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Θέλουμε τις πιο ψηλέ προδιαγραφές και πρότυπα, την προστασία της ειρήνης στη Βόρεια Ελλανδία και το δημοκρατικό έλεγχο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Όλα τα υπόλοιπα ε, της ε, ε, εντολής τα βλέπουμε επικριτικά μέχρι και απορριπτικά. Η συνεργασία μυστικών υπηρεσιών, η στρατιωτική συνεργασία στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Εμείς θέλουμε η δική μας ε, ε, πολίτες ε, να γνωρίζουν τα πράγματα και να ξέρουν ότι δεν έχει αποτραπεί ακόμα το σκληρό Brexit, το άτακτο. Χάνσεν για 1,5 λεπτό. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά τη μεταβατική φάση, το κόστος του Brexit θα έχει ξεπεράσει ε, το σύνολο των εισφορών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση από τότε που εντάχθηκε πριν από 47 χρόνια. Είναι πραγματική τρέλα από πλευράς οικονομικής και δικαιώνονται όσοι το πιστεύουν αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον στις πόρτες Ευρωπαϊκής Ένωσης μία από τις πιο δυναμικές οικονομίες. Ε, από πλευρά διεθνού εμπορίου πρέπει να πω ότι αυτό που προσφέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ περισσότερο από όλες τις άλλες συμφωνίες. Ε, σχέση χωρίς ποσοστώσεις, χωρίς θελωνιακούς δασμούς. Αυτό ζητάει από την άλλη ε, θεμητό και ίσο ανταγωνισμό για να μην έχουμε ε, dumping κοινωνικό, περιβαλλοντικό, φορολογικό και κανονιστικό. Αυτό που ονομάζουμε ισότιμους κανόνες ε, παιχνιδιού θα πρέπει να είναι αντίστοιχο της πρώτης εθνικής ποδοσφαίρου στην Αγγλία, της Premier League. Θα πρέπει να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Όταν πρόκειται για ευρωπαϊκό δίκαιο, ε, το τελεσίδικο όργανο θα πρέπει να είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μπορεί το ελεύθερο εμπόριο ποτέ να υποκαταστήσει την ε, ιδιότητα του μέλους. Είναι πολύ περιοριστικό κατά τέτοιο το χρονοδιάγραμμα που επιβάλλουν οι Βρετανοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η Πρόεδρος. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τώρα θα δώσουμε ε, το λόγο ε, στον κύριο Σίλβα Περέρα και χαιρετίζω τους πολίτες που μας ακούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα όσον αφορά τι πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμέ για τι διαπραγματεύσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. 21 σελίδε, 103 παράγραφοι. Αλλά θα έλεγα ότι ίσω το πιο σημαντικό είναι η πρώτη σελίδα. Το εξώφυλλο που έχουμε ουσιαστικά τι υπογραφέ των επικεφαλής των βασικών πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που είναι υπέρ αυτού του ψηφίσματος και δείχνει ουσιαστικά ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι στο να προασπίσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και το κοινό μας όραμα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνουμε και έκκληση προς τα κράτη-μέλη να πράξουν ακριβώς το ίδιο. Να αρνηθούν οποιασδήποτε διμερείς διαπραγματεύσεις στο επίπεδο αυτό και να λειτουργήσουν από κοινού με νέα φωνή μέσω της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω του επικεφαλή διαπραγματευτή και μοναδικού διαπραγματευτή του κυρίου Μπαρνιέ. Είμαστε σαφεί για το τι θέλουμε να πετύχουμε μια φιλόδοξη στρατηγική πολιτική οικονομική σχέση με το Μένο Βασίλειο. Παράλληλα όμως λέμε ξεκάθαρα και ηχηρά ότι θέλουμε να έχουμε έναν ανοιχτό αλλά και ισότιμο θεμητό ανταγωνισμό, ισοτιμία στις σχέσεις, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και καμία υποχώρηση όσον αφορά τα υψηλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια καμία υποχώρηση όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στέλνουμε επίση μέσω του ψηφίσματος αυτού και κάποια μηνύματα. Και έχουμε δει ότι υπάρχει και μία ανταπόκριση αρνητική από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την ε, μετέπειτα πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ουσιαστικά θα υποβαθμίσει τη μελλοντική εμπορική συμφωνία. Α μην ξεχνάμε επίση ότι ο πρώτο πυλώνα ε, τη μελλοντική οικονομική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχει συμφωνηθεί στα πλαίσια τη Συμφωνία Αποχώρηση ε, και έχει να κάνει βασικά με τη Βόρεια Ιρλανδία. Η ευθυγράμμιση που, για τους κανόνες της Βόρειας Ιρλανδίας και η συνοριακή έλεγχη στην θάλασσα της Ιρλανδίας. Θα επεξεργαστούμε λοιπόν μια μελλοντική συμφωνία, αλλά θέλουμε επίση να εφαρμόζονται πλήρω οι δεσμεύσει που ήδη υπάρχουν στα πλαίσια τη συμφωνία αποχώρηση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Πέτερσεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια λυπηρή ημέρα όταν μια τόσο μεγάλη χώρα ε, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εκείνους και για εμάς. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αποτελεί πολύ θετικό το γεγονός ότι το ψήφισμα που συζητούμε σήμερα είναι τόσο ολοκληρωμένο και έχει συνταχθεί με τόσο ευρεία υποστήριξη από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί αυτό αποστέλει και ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα, ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε ένα σύνολο δίκαιων κανόνων για τις μελλοντικέ μας σχέσεις και τη μελλοντική μας συνεργασία. Γιατί γιατί δεν είναι καλό να ανταγωνιστούμε σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικά, εργασιακά, καταναλωτικά, ούτε να ανταγωνιστούμε για το ποιο έχει του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστές. Ούτε ε, μπορούν όλα αυτά ε, να σημαίνουν ότι η, Ευρωπαϊκή, ε, ε, η Βρετανία θα έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να τηρεί συγκεκριμένε υποχρεώσεις και πρότυπα. Θέλουμε να διατηρήσουμε βεβαίως την ενιαία αγορά. Είναι το πιο σημαντικό η πιο σημαντική κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω, θα αντιμετωπίσουμε πολλέ προκλήσει όσον αφορά την αλεία. Υπάρχουν πάρα πολλέ θέσει εργασία που διακυβεύονται, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και ζουν από την αλληλεία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι μελλοντικέ ε, αλληλευτικές συμφωνίες να μην ε, αποτελέσουν ξεχωριστό αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όλα θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολε αυτές οι διαπραγματεύσεις σε ένα δύσκολο περιβάλλον, αλλά στόχο ε, νομίζω ότι πρέπει να είναι να καταλήξουμε σε μια συνεργασία η οποία θα είναι ισχυρή για όλου. Ευχαριστώ. Και το λόγο έχει ο κύριος Νικολαμπή. Όντω, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να έχουμε προνομιακή σχέση με τον Μένο Βασίλειο. Είναι, είμαστε πάρα πολύ κοντά όσον αφορά την οικονομία και τον πολιτισμό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μόνο εκχωρήσει προ τον Μένο Βασίλειο. Ο κύριο Μπαρνιέ μα είπε ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε όλε τι ποσοστώσει και όλου του δασμού, τι ανταλλαγέ που θα έχουμε με τον Μένο Βασίλειο. Άρα, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών πλήρη. Την ίδια πρόταση έκανε και ο κύριο Λάμπερ πριν από λίγο. Συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών συνάπτουμε μόνο τον κόσμο, σε λίγο και με το Βιετνάμ. Από την άλλη όμως δεν δεχόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει στην Τελωνιακή Ένωση. Είναι τρίτη χώρα και επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώ ποια προϊόντα φτάνουν στην χώρα αυτή και αν μπαίνουν χωρί ελέγχου τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α προστατεύσουμε συγκεκριμένου τομεί όπω του Γάλλου Αλεί, οι οποίοι ένα 30% του κύκλου εργασιών του το πραγματοποιούν στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά μέσω του τομέα τη έχουμε ένα εργαλείο μόχλευση πάρα πολύ σημαντικό σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι υπάρχουν και οι ιδέες του Πρόεδρου Τραμπ, τον οποίο δεν εκτιμάται καθόλου και οι οποίες όμως λειτουργούν όσον αφορά το τομέα της οικονομίας. Νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε αυτή τη στιγμή μέσω του Brexit να αλλάξουμε και εμείς το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε στην οικονομία και να το εφαρμόσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντια έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Είναι ιδιαίτερη στιγμή αυτή γιατί είναι η πρώτη φορά που συζητάμε εδώ στο Brexit στο Κοινοβούλιο χωρίς να είναι οι Βρετανοί συνάδελφοί μας εδώ και πρέπει να πω ότι εκτός από μια ομάδα που ήταν εκεί πάνω πραγματικά μου λείπουν πολύ και νομίζω ότι αυτό δείχνει πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι έγινε αυτό το Brexit. Είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να κάνω ε, ε, το εράσμους μου στην, στο Εδιμβούργο. Ακόμα και όταν, σήμερα όταν πηγαίνω εκεί νιώθω ότι είναι το σπίτι μου και αυτό και νομίζω ότι αυτές τις αναμνήσεις πρέπει να τιμήσουμε και στο μέλλον. Και οι οικονομικές και εμπορικέ μας σχέσεις βεβαίως θα είναι ζωτική σημασία για το μέλλον. Όμως αν θέλουμε γερά θεμέλια στη σχέση μας πρέπει να, να δούμε και άλλα ζητήματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πρόγραμμα Εράσμους. Οι νέοι δεν ψήφισαν υπέρ του Brexit και νομίζω θα ήταν σφάλμα να να στερήσουμε τις, τις ευκαιρίες από τα παιδιά αυτά, από τους νέους αυτούς ε, που είχαμε εγώ και πολλοί συνομήλικοί μου. Γι' αυτό και πρέπει να, χρειάζεται, να οικοδομήσουμε μια στενή συνεργασία και μέσω του προγράμματος ε, Εράσμους, ώστε να διατηρηθούν οι γέφυρες για να μπορέσουν οι Βρετανοί να γυρίσουν στο σπίτι τους. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ως CCR υποστηρίζουμε το ε, ψήφισμα αυτό. Ανησυχητικό όμως είναι το πνεύμα που επικρατεί ε, στη συζήτηση και στι διαπραγματεύσει. Η ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ Βρυξελών και Λονδίνου δεν μας κάνει αισιόδοξου. και είναι προφανές ότι ένα, μια τρίτη χώρα βεβαίως δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με τα, με τα ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη-μέλη του ΕΟΧ ή του ΕΦΤΑ. Όμως ε, η Βρετανία θα παραμείνει ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έχει πολλούς δεσμούς με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ιστορικούς δεσμούς, κοινωνικούς δεσμούς, οικονομικούς δεσμούς. Ακόμα και στις πιο σκοτεινές σελίδε της ιστορίας μας, Ακόμα και το 1945 η Μεγάλη Βρετανία ε, βεβαίως επέδειξε ηρωισμό και ε, υπερασπίστηκε τις ευρωπαϊκές αξίες όπως και η Πολωνοί. Γι' αυτό και είναι κοινό μας συμφέρον να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες ε, σχέσεις. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν ποτέ οι διαπραγματευτές μας. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βιλανουέβα Ρουίθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έξοδο του, Ινω... του Ηνωμένου Βασιλείου μα ανοίγει ένα παράθυρο για να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντε και να μην τα επαναλάβουμε. Ρητορική μίσου, ε, αβεβαιότητα, ανασφάλεια. Θα πρέπει να τερματιστεί. Θα πρέπει να είναι πρόοδο και αλληλεγγύη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, δεν μπορούμε να ποντάρουμε στην απογοήτευση και σε αποτυχημένα εγχειρήματα που διώχνουν τον κόσμο. Θα πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα του κόσμου, των πολιτών που ζουν 140.000 περίπου Ισπανοί ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μα ανησυχεί η κατάσταση των εργαζομένων. 15.000 κάθε μέρα περνούν τα σύνορα του Γιβραλτάρ. Η κατάστασή του ακόμα είναι αβέβαιη. Θα πρέπει να αγωνιστούμε αποφασιστικά κατά του κοινωνικού και του φορολογικού ντάμπινγκ. Διαφωνούμε με μεγάλο τμήμα ε, τη διαπραγματευτική εντολή για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και να πάμε σε θέσει πολύ πιο προληπτικέ των συγκρούσεων και των σειράξεων και να μην πληρώνουν τα σπασμένα πάντα οι λαοί. Η δική μα πολιτική ομάδα θα συνεχίζει να θωρακίζει τα δικαιώματα των πολιτών, τα περιβαλλοντικά του πρωτογενού τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, για να μην ρημάζει η πεθρό και τα χωριά μα. και να μην είμαστε ένα αντάλλαγμα για άλλα συμφέροντα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταγιάννη, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, το κείμενο το οποίο θα ψηφίσουμε έχει ως στόχο να ενισχύσει την ενότητα μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποστηρίξει στεναρά τον Μισελ Μπαρνιέ για να υποστηρίξει τη βασική διαπραγματευτική μας θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περασπίσουμε την εσωτερική μας αγορά. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην εσωτερική αυτή αγορά σαν δούριο ύπο χωρί να σέβεται πραγματικά πρότυπα και κανόνε. Και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε ουσιαστικά να προστατεύσουμε επιχειρήσει και του Ευρωπαίου πολίτε. Η υγεία επίση των πολιτών θα πρέπει να διασφαλίζεται έτσι ώστε τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν πραγματικά να σέβονται τα δικά μα τα πρότυπα και σε καμία περίπτωση να μην βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εμεί θέλουμε να τρώμε παρμεζάνα στην Ιταλία και όχι πάρμεζανα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να καταφέρουμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και στα έγγραφα στο διαδίκτυο και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να, τον, να προστατεύσουμε όλου του τομεί όπω τον τομέα τη ενέργεια, τη βιομηχανία και βέβαια να προστατεύσουμε του πολίτε που βρίσκονται στην Ιρλανδία και στο Γεβραλτάρ. Από κοινού να αντιμετωπίσουμε και τι προκλήσει τη τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει το Ηνωμένο να γίνει μια Σιγκαπούρη στι όχθε μα, τόσο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε το δυνατόν πιο θετικέ σχέσει με το Λονδίνο, το οποίο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παραμένει ουσιαστικά ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Λάγκε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ψήφισμα καταδεικνύει ότι είμαστε έτοιμοι ε, να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε εντός ε, εννέα μηνών να οργανώσουμε μια τέτοια ε, συμφωνία εμπορική. Γιατί η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Συνήθω έχουμε δύο διαφορετικούς εταίρους που κάπως προσεγγίζουν ένα τον άλλον, γίνονται κάποιες συνονοήσεις, επαφέ για κοινά πρότυπα, αναγνωρίζονται τα πρότυπα του ενό από τον άλλον κτλ. κτλ. Τώρα όμω έχουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα και θέλουμε να αποφασίσουμε πόσο μπορούμε να αποκλίνουμε. Από αυτή την άποψη είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, λίγο πιο άνετα από τι άλλε διαπραγματεύσει. Γιατί συνήθω ε, πρέπει να, Γιατί όπω και πάντα πρέπει να ε, ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι πυλώνε. Βεβαίω, ε, κατάργηση δασμών. Αυτό είναι ένα εφικτό στόχο. Βεβαίω, πρέπει τα προϊόντα τα βρετανικά που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πραγματικά βρετανικά και όχι προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη Βρετανία. Δεύτερον, Ζητούμενο είναι τα πρότυπα των προϊόντων και των ε, υπηρεσιών. Εδώ υπάρχει ένας σαφές ε, σύνολο κανόνων όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, την προστασία της δημόσιας υγείας, τα πρότυπα δεν μπορούν αυτά να αμφισβητηθούν πουθενά. Και σε αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι οι συνεννοήσει θα είναι σχετικά εύκολε. Ο τρίτο πυλώνα είναι ο πιο περίπλοκο. Φυσικά υπάρχουν και οι κανόνε που διέπουν το εμπόριο ώστε να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Όπως για παράδειγμα το ζήτημα ίσων δικαιωμάτων στην εργασία, ε, ίσα περιβαλλοντικά πρότυπα ίσα, ε, ίσοι κανόνε όσον αφορά τι επιδοτήσει, κρατικέ ενισχύσει και το ζήτημα ε, ενό εναρμονισμένου φορολογικού συντελεστή. Διότι διαφορετικά θα είχαμε στρέβλωση του ανταγωνισμού και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Όταν, αν υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού, τότε βεβαίω και θα πρέπει να εισαγάγουμε δασμού για να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε την κατάσταση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο στη διαπραγμάτευση αυτή ότι θα υπάρχει ένα, μια, ένα νησί μετά, ε, από την απέναντι πλευρά της μάχης η οποία στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ο κύριος Γκαρικάνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπαρνιέ για το έργο σας και τις προσπάθειές σας. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή σχέσεων, ελπίζω να είναι γόνιμη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα ήθελα να στείλω ένα σαφέστατο μήνυμα προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το κοινοβούλιο μας δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει το Ηνωμένο Βασίλειο φορολογικός παράδεισος ή πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος έξω από την Ευρώπη, στις όχθες μας. Θυμίζω ότι παράγραφο 21 του ψηφίσματος λέγει «Πιστεύουμε σε ότι το, Ευρωπα... το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συμμετέχει στην ε, νομοθεσία κατά του ξεπλήματος ε, με ανταλλαγή πληροφοριών, με διαφάνεια των τραπεζών και μέτρα ε, κατά του φορολογικού dumping. Και αυτό ισχύει και για τη Βερμούδα, το Καϊμάν, τις Παρθένους νήσους και όλους ε, τους άλλους ε, τόπους που έχουν χαμηλή ε, φορολογία καταθέσεων ή επιχειρήσεων. Ε, κύριε Μπαρνιέ, αυτό το ζήτημα είναι υπαρξιακό για την Ευρώπη. Αν επιτρέψουμε φόρο διαφυγή, φόρο ε, αποφυγή στα ανοιχτά της Ευρώπης, κινδυνεύει ο πληθυσμός μας. Αυτό θα πρέπει να είναι μία από τις υψηλότερες, για να μην πω υπαριθμών ένα, προτεραιότητα. Ο κύριος Καμπενώση, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα υψηλό βαθμό υποκρισία εδώ. Θα ψηφίσουμε αύριο αυτό το σχέδιο ψηφίσματο. Μπορεί να έχει κάποια θετικά στοιχεία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ρίχνουμε αυτή τη στιγμή κροκοδίλια δάκρυα για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουμε λίγο μια στάση λίγο σχιζοφρενική, θα έλεγα ακόμα και στα λόγια της ε, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλάει για φίλους, φίλους κτλ. Ενώ εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια, αντί να αναλωνόμαστε σε τόσε πολλέ δηλώσει, θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από το να θελοτυφλούμε και να λέμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να φύγει ποτέ και ότι κάνανε λάθο οι, Ευρωπαίοι, οι Βρετανοί πολίτε και το καθεξής. Μιλάμε επίση για όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία θα ψηφίσουμε αύριο και θα πρέπει να διέπουν την μελλοντική μα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχάς να δείτε ότι κυρίως τα προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτά τα οποία θα πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι τόσο πολύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά θα πληγεί πάρα πολύ ο δικός μας παραγωγικός τομέας. Ο κύριος Μπούρζουα, παρακαλώ, από την ομάδα Σιάρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, έχει έρθει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει γρήγορα και λογικά, ρεαλιστικά, αλλά ταυτόχρονα να ε, προχωρήσει σύμφωνα με την πολύ ευρεία διαπραγματευτική εντολή. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο Μισελ Παρνιέ με τις εξαιρετικές επιδόσεις του μέχρι τώρα. Τώρα θα πρέπει να έχουμε μια εμπορική συμφωνία χωρίς φραγμούς, συνολική, που να σέβεται τις κόκκινες γραμμές μας να έχουμε ισότιμους κανόνες παιχνιδιού αλλά και μια πολύ καλή συμφωνία, μια περισσότερη ασφάλεια, ε, αλληλεία, άμυνα κτλ. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να μας απαντήσει. θα συνεργαστεί ε, στην συνεργασία την ενεργειακή της Βόρειας Θάλασσας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον 21ο αιώνα χρειαζόμαστε πιο εντατική συνεργασία για τη λεγόμενη γαλάζια, θαλάσσια οικονομία. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση των Οκεανών. Ευχαριστώ ο κύριος Σόλτς από την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε όλοι έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν πολλά σημαντικά στη ε, σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο που πρέπει τώρα να ρυθμιστούν. Αυτό είναι το καθήκον μας υπέρ των πολιτών μας στα κοινωνικά, ε, οικονομικά, οικολογικά και πολιτιστικά θέματα. Άρα είναι λιγότερο μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών και περισσότερο για δίκαιες ε, εμπορικές σχέσεις χωρίς αποκλεισμούς. Το θεωρώ αμφίβολης ε, σκοπιμότητας να κάνουμε ε, ό,τι με το TTIP, ε, όπου να τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, και τα αμυντικά και τα αστυνομικά και τα υπόλοιπα, που να διαφεύγουν του κοινοβουλευτικού ελέγχου και να απαντούν σε αυτά και να αποφασίζουν κάποιες εξωτερικές επιτροπές. Ζητώ από το Συμβούλιο να δημιουργήσετε σαφήνεια με δημοκρατικό τρόπο. Υπάρχουν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης ε, του ΟΗΕ, η Συμφωνία των Παρισιών, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μην κάνετε εκπτώσεις στις φιλοδοξίες που έχουμε για το περιβάλλον και την ασφάλεια των προϊόντων, ε, θεωρώντας αυτά τα θέματα εμπορικής σημασίας. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Γκοζάλης Πόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν Κάποιο οργανώνει ένα Brexit είναι για να φύγει, όχι για να μείνει φεύγοντα. Δεν μπορεί να έχει περισσότερα πλέον εκτήματα το ΕΒ Βασίλειο όντα απ' έξω από εκείνα που είχε όταν ήταν μέσα. Τρία χρόνια κλεγόμαστε που φύγανε. Ε, τώρα δεν μπορεί να μα πιάσει η νοσταλγία που μα έφυγαν. Ε, τώρα είναι τρίτη χώρα. Α διαπραγματευτούμε σκληρά, όπω το κάνουμε με κάθε τρίτη χώρα. Και α υπερασπίσουμε του δικού μα την αποαπικιοποίηση του Γιβραλτάρ που δεν θα πρέπει να γίνει φορολογικός παράδεισος ή να παραμείνει. Ας υπερασπιστούμε τους ψαράδες μας που καθημερινά θαλασσοπνίγονται για να βγάλουν το ψωμί τους. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους αγρότες μας, τα προϊόντα μας. Αν εκείνοι οι Βρετανοί πολίτες και πολιτικοί θέλησαν να είναι τρίτη χώρα, ας τους φερθούμε ως αυτό που είναι τρίτη χώρα. Έχει φύγει από, το Ηνωμένο, από την Ευρώπη το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν πρέπει να γίνει μια νέα νότιο-ανατολική Ασία μπροστά από την πόρτα μας. Συγγνώμη κύριε Πέτερσεν, νομίζω ότι έχετε ε, το flash στο κινητό σας αναμένω. Μπορείτε να το σβήσετε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θέσει τις δικές του προτεραιότητες για τις ε, μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορούμε να επιτύχουμε μια συμφωνία στο τέλο του έτους και τι είδου συμφωνίε θα είναι. Φυσικά ένα, μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με ένα κράτος μέλος και φυσικά οι διαπραγματεύσει πρέπει να βασίζονται στις τέσσερις ελευθερίες, την ευημερία και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό βεβαίω θα είναι αποφασιστική σημασία. Ιδίω στην εξωτερική πολιτική για άμυνα, ελπίζω το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και του ΝΑΤΟ να συνεχίζει να συμμερίζεται τις δικές μας ε, αξίες. Στην, σε επιχειρήσεις, σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων, ε, στην περίπτωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, του αφοπλισμού, του πυρηνικού αφοπλισμού, Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει ενότητα εν ώψη των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τους Βρετανούς συναδέλφου για την εξαιρετική συνεισφορά τους ε, στα ευρωπαϊκά πρότυπα που βελτίωσαν συνολικά τη ζωή και το επίπεδο διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σραίνεμαχα. Η κυρία Σχρένεμακερ, έχει έρθει η ώρα να χτίσουμε το μέλλον μας με τους Βρετανούς συναδέλφους. Ας δούμε το κοινό συμφέρον και τους στόχους μας και πώς θα το εξυπηρετήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην κοιτάμε μόνο αυτά που μας χωρίζουν. Γι' αυτό επιμένω σε μια φιλόδοξη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που να δημιουργεί τα θεμέλια για σωστό και δίκαιο ανταγωνισμό. Τούτων λεχθέντων, μια τρίτη χώρα προφανώ δεν μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια προνόμια με ένα κράτο μέλο τη Ένωση και τα ίδια ωφέλη ανοιχτή η αγορά μας, αλλά θα πρέπει αυτό να συνδυάζεται με την προθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να προσαρμοστεί και να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες και τα πρότυπά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη, να διατηρήσουμε ψηλά τα πρότυπά μας και τους κανόνες μας για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό και να αγωνιστούμε πριν το καλοκαίρι να υπάρχει συμφωνία για την αλία. Λυπάμαι για τον Brexit και θα συνεχίσω να λυπάμαι, αλλά τώρα θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και να χτίσουμε νέα σχέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ντέιβιτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φοβούμε ότι πολλοί υποστηρικτές ε, μιας Ευρώπης χωρίς σύνορα νιώθουν συναισθήματα εκδίκησης. Υπόθηκε ότι η, Βρετανία δεν θα πρέπει να έχει την αυτονομία να αποφασίζει για τις δικές της ε, υποθέσεις. Όμω η Βρετανία είναι μέλος του ΠΟΕ και η Ευρώπη δεν μπορεί εδώ να δημιουργήσει τεχνητά εμπόδια. Έχουμε μεταφορές, έχουμε γεωργία, ναι όλα αυτά ισχύουν, αλλά στην εποχή του ίντερνετ δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί τεχνητά εμπόδια, για παράδειγμα στις, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ε, Βρετανίας, ούτε μπορεί κανείς να ε, ε επηρεάσει αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έκανε με κυρώσεις, όπως έκανε η Ρωσία η οποία ε, εν πάση περιπτώσει κατάφερε και πέτυχε την ε, αυτάρκειά της μέσα σε δύο χρόνια μετά την επαβολή κυρώσεων. Όλα αυτά τελικά θα πλήξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα την ωφελήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουχαδέ. Ευχαριστώ. Ε, τέλειωσε το τσίρκο του, εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Λέσχη. Τώρα θα πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά για οικονομικέ και εμπορικέ συμφωνίε που να εγγυώνται τα δικαιώματα των δικών μα πολιτών. Α πούμε, οι Ισπανοί πολίτε να μπορούν να ψαρεύουν οι αλήθεια εκεί. Η ελεύθερος ανταγωνισμός των ε, γεωργικών προϊόντων, αλλά και σε θέματα όπω είναι η ασφάλεια ή η δικαστική συνεργασία. Α διαπραγματευτούμε σκληρά και όχι λιγότερο σκληρά από ό,τι κάνουμε με τρίτες χώρες με τις οποίες συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίες. Υπό την έννοια αυτή έχει έρθει η ώρα για να τερματίσουμε με την ιστορία του Γιβραλτάρ, να τελειώσει αυτή η απικιοκρατικοποίηση, να σταματήσει αυτή η ε, βρετανική απικία, ε, η παρασιτική, με τον αθέμητο ανταγωνισμό σε ισπανικό έδαφος. Το Γιβραλτάρ έχει γίνει πλυντήριο χρήματος από εγκληματικέ δραστηριότητες, εκεί νομιμοποιούν τα έσοδά του. Θα πρέπει να βάλετε τα θεμέλια στην Κομισιόν για να σπάσει, τελειώσει αυτή η απικία. Το ξέρουμε ότι είναι ευθύνη της ισπανικής κυβέρνησης, αλλά σε αυτή τη λέσχη που είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς εταίροι θα πρέπει να έχουμε αντίστοιχες απαιτήσει για συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Χιούμπνερ. But... Ένα λεπτό. Συγγνώμη, δεν, δεν ξέρω αν είδατε τον κύριο Φλ... Δεν είδα τον κύριο Φλάναγκαν, με συγχωρείτε. Oh, sorry, at the catch the eye, I'll give you the floor. Στη διαδικασία Catch θα σας δώσω το λόγο. Συγγνώμη. Κυρία Χιούμνερ, έχετε το λόγο. Thank you for the second chance. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία να πάρω το λόγο. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη μελλοντική σχέση που θα έχουμε με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρουμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα έχει ένα πολύ μικρό κεφάλαιο όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές αυτές υπηρεσίες και θα προβλέπονται μόνο κάποιες εξαιρέσεις και κάποιες αποκλήσεις. Θα υπάρχουν επίσης κάποιοι μηχανισμοί ισοτιμίας για να έχουμε μία σχέση με το Μένο Βασίλειο στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ελάχιστους μήνες στη διάθεσή της προκειμένου να δημιουργήσει αυτούς τους μηχανισμούς ανταπόκρισης και θα έχουμε ελάχιστο χρόνο για να καταφέρουμε τελικά να προσαρμοστούμε. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το πλαίσιο ισοτιμίας προκειμένου να μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό με το Μένο Βασίλειο. Πρόκειται όμω για ένα αυθαίρετο τελικά εργαλείο, το οποίο για να λειτουργήσει στην πράξη θα χρειαζόμαστε επικοδομητική συνεργασία με του Βρετανού ρυθμιστέ, προκειμένου να έχουμε ακαιρεότητα στη δική μα τη χρηματοπιστωτική οικονομική αγορά και να μπορούμε να προστατεύουμε του Ευρωπαίου πολίτε, καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια φιλόδοξη και επιτυχή μελλοντική σχέση με το Μένο Βασίλειο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει το συντομότερο δυνατό και εμεί να ολοκληρώσουμε την τραπεζική μα ένωση και να δημιουργήσουμε πραγματική ένωση κεφαλαιαγορών. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε αποτελεσματική επιτήρηση, αλλά αποτελεσματική επιτήρηση έχει και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα τη Αγγλία έκανε συγκεκριμένε δηλώσει όσον αφορά το σύστημα επιτήρηση και παρακολούθηση. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει και εδώ πέρα να υπάρχουν ισότιμοι κανόνε. Σα ευχαριστώ. ο κύριο ε, Ντακάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από τις ε, πιο σκοτεινές αυτές, αν θέλετε, σελίδες που είδαμε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας δίνεται επιτέλους η ευκαιρία να καταφέρουμε τελικά να διασώσουμε τα 25 αυτά χρόνια ευρωπαϊκής οικοδόμησης για τους Ευρωπαίους πολίτες, προσπαθώντας να έχουμε ισότιμα πρότυπα με το Μένο Βασίλειο στον αφορά το κοινωνικό τομέα, τον περιβαλλοντικό τομέα και το φορολογικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε εμεί τα πρότυπα της παραγωγής, τα πρότυπα της ασφάλειας των τροφίμων δεν θα πρέπει το Ενωμένο Βασίλειο να λειτουργήσει ω δούριος ύπο και κατά αυτόν τον τρόπο να εισαχθούν στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκής Ένωσης τρόφιμα τα οποία θα ήταν ε, επιζήμια για την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και επιζήμια από οικονομικής πλευράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσει. Α μην ξεχνάμε επίση ότι έχουμε κοινού πολιτικού δεσμού, πολιτισμικού δεσμού με το Ενωμένο Βασίλειο και οι πολιτισμικοί αυτοί δεσμοί έχουν να κάνουν ακόμα και με την κοινή αγροδιατροφική παραγωγή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει και αυτόν το προασπίσουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι μετά το Brexit δεν θα προκύψει ένα τεράστιο κενό, αλλά μια Ευρώπη η οποία θα είναι συνεχώ πιο ισχυρή και πιο βιώσιμη και θα είναι έτοιμη να προασπίσει όλο και περισσότερο του πολίτε τη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντρους έχει το λόγο. Με μεικτά συναισθήματα παρεμβαίνω εδώ πρώτη φορά σε